Fine, Να αρχίσουμε. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση αυτής. Η κυρία Λούλινγκ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι στην ημερήσια διάταξη την αυριανή έχει την ψηφοφορία για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, στη ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για μια έκθεση που σκοπό έχει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροποποίηση των κειμένων για τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις μας παρουσίασε το κείμενό της επί του θέματος αυτού. Την περασμένη εβδομάδα και έχουν οριστεί ήδη και οι Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Συνεχίζουμε μια διαδικασία που δεν ε, χρησιμεύει ε, σε τίποτα. Θα ήταν λίγο περίεργο να συζητήσουμε τέλη Οκτωβρίου τις συστάσεις αυτές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, την ε, κατάρτιση των κειμένων αυτών, ενώ τα κείμενα ήδη τα έχουμε στη διάθεσή μας. Τι να σας πω. Εγώ προτείνω αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, να το βγάλουμε από την ημερήσια διάταξη, γιατί τι να σας πω, είναι σαν ε, αναμασιμένο πιάτο. Εφόσον έχουν οριστεί οι εισηγητές για τις δικές μας προτάσεις επί των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο Φιλίπ. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω τα σχόλια της Astrid Gluling και πριν από μερικούς μήνες το είχα πει και εγώ. Ε, αν έχει νόημα δηλαδή μία έκθεση μετά την ε, δημοσίευση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε είχε νόημα τότε θα ήταν η σωστή χρονική στιγμή να το σταματήσουμε. Όμως ε, αφιερώσαμε πολύ ενέργεια και κάναμε πολλή δουλειά για το θέμα αυτό. Έχουμε μια έκθεση που όντω ε, μπορεί να βελτιώσει τις προτάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε προτείνω τελικά όντω να το ψηφίσουμε αύριο, να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, να το ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ καθυστερημένο και σε κάποιο βαθμό όντω ε, ε, έχει καθυστερήσει. Και δείχνει τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ε, τα ε, νομοθετικά αυτά κείμενα. Οπότε εγώ προτείνω να το ψηφίσουμε αύριο, να το ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια και να ε, τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Η κυρία Λούλινγκ θέλει πάλι να πάρει το λόγο. Όταν συζητήσαμε τις τροπολογίες την περασμένη εβδομάδα μας είπαν ότι θα υπήρχαν συμβιβαστικές τροπολογίες. Εγώ ήθελα να τις μελετήσω κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν τι έχω. πώ μπορώ να ψηφίσω αύριο το πρωί για τροπολογίε συμβιβαστικέ που δεν τι γνωρίζω ακόμη. Κοιτάξτε, είναι μία ε, μέθοδος εργασίας ε, που δεν είναι σοβαρή. Και θα ήθελα να το πω ε, και στο συνάδελφό μου. Εγώ 25 χρόνια ήμουνα σε Εθνικό Κοινοβούλιο και ποτέ δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο. Να ψηφίσουμε συστάσεις προς τις κυβερνήσεις, ενώ τα κείμενα των κυβερνήσεων έχουν ήδη κατατεθεί. Ε, νομίζω. Μάλιστα. Κυρία Λούλινγκ, το Προεδρείο γνωρίζει το γεγονός αυτό, ότι έχουμε κάπως, ε, μας έχουν προλάβει εξελίξει. Είναι κάτι όμως που το γνωρίζαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και η ομάδα εργασίας ε, του Προέδρου ε, Φαν Ρόμπαϊ εξετάζει το ζήτημα αυτό και αποφασίσανε ότι τα στοιχεία που ε, συνιστούν αλληλεπικάλυψη με, τα, με, τις επιτρο, με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρησιμεύσουν ως καθοδήγηση στο νομοθετικό αυτό πλαίσιο. Δεν λέω βέβαια ότι όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρονται στο έγγραφο στις, ε, στην έκθεση στην έκθεση ΦΕΟ θα ληφθούν υπόψη. Και από ό,τι κατάλαβα, ε, προτείνει και η ίδια ε, και η έκθεση νέε τροπολογίε επί, την, ε, επί της εκθέσεως για να βελτιωθεί το κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το, αυτή η μερική ε, αλληλεπικάλυψη δεν είναι πλήρης τελικά. Κυρία Λούλινγκ, κοιτάξτε, τότε θα πρέπει να δώσουμε λίγο στον εισηγητή το χρόνο να αναθεωρήσει το κείμενό του και να δούμε κατά πόσο ε, καταλήγουμε σε κάτι που έχει νόημα να το ψηφίσουμε και που στέκει ως κείμενο. Ίσως να μπορέσουμε να το αναβάλουμε σε, για, δύο, για εβδομάδες για να έχουμε χρόνο ε, να το ε, ελέγξουμε. Δεν νομίζω ότι είναι ε, Προ τιμή μα αυτό το πράγμα. Δεν φαινόμαστε σοβαροί έτσι. Και εγώ πολλά χρόνια ήμουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Um, Νομίζω ότι καλό θα ήταν οι εισηγητές των πολιτικών ομάδων θα έπρεπε να το εξετάσουν αυτό, οι συντονιστές να το εξετάσουν ε, πώς ε, θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν και προφορικές τροπολογίες που έχουν προγραμματιστεί. Η κυρία Λούλινγκ λέει να αναβάλουμε την ψηφοφορία, αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι για να μην γίνει αυτό. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές να εξετάσουν τις προφορικές τροπολογίες του κυρίου Φέιο, ώστε να μην καθυστερούμε την ψηφοφορία του συγκεκριμένου κειμένου. Υπάρχουν άλλα σχόλια? Would Κύριε Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ξαναφύγω διότι διαπραγματεύομαι με την Προεδρία και το Συμβούλιο την ε, ακριβή, ε, την ακριβή διατύπωση του, της οδηγίας ε, IFM αλλά νομίζω ότι η έκθεση Φέγιο ήταν μια δουλειά σωστή η οποία προχώρησε καλά υπάρχουν συμφωνίες και δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη σειρά μας με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε δεν μπορώ να κάνω τρία πράγματα μαζί θα επανέλθω Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Στην περίπτωση αυτή θα προχωρήσουμε. Εκτός και αν θέλετε να ψηφίσετε. Κυρία Λούλινγκ. Προφανώς οι άλλες ομάδες πρέπει να ξέρουν τι θα γίνει. Δηλαδή αυτοί που δεν ε, ήταν εδώ, εγώ παρουσίασα το πρόβλημα και είπα ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι η έκθεση αυτή ε, ε, είναι ακόμη σε πολύ συγκεχημένη κατάσταση και θέλει βελτίωση και ε, ξαναχτένισμα και δεύτερον οι συγητές που είχαν το κείμενο πρέπει να έχουν χρόνο εγώ Θέλω να βλέπω τα κείμενα. Ακόμη και αν έχω τεράστια εμπιστοσύνη στο συντονιστή μου, θέλω να δω τα κείμενα και οι συμβασικές τροπολογίες που μας ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα δεν είναι ακόμη διαθέσιμες τώρα δεν επιπλέον ε, δεν μπορούμε καν να, ε, ε, να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και προφορικές τροπολογίες που μας ανακοινώνουν. Πώς λοιπόν θα ψηφίσουμε αύριο στις 10.30 το πρωί, δεν είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά νομίζω ότι ο πιο εμπλεκόμενος θα είναι ο κύριος Φέγιο. θα φτάσει αλλά έχει πρόβλημα αεροπλάνου. Προχθές ήταν το τρένο, τώρα είναι το αεροπλάνο. Παρακαλώ λοιπόν κάντε λίγο υπομονή και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά λογικό και προφανώς οι συντονιστές θα ενημερωθούν για τη θέση σας και φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουν μετά από αυτή τη συνεδρίαση. Έχω ορισμένες ανακοινώσεις εν ονόματι της Προεδρίας. Το πρώτο είναι η συμμετοχή την 1η ε, ε, Σεπτεμβρίου ναι, ε, ε, για την, ε, στη συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ. Ένας εκπρόσωπός μας υπήρξε στη συνάντηση αυτή και παρουσιάστηκε η κατάσταση και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και υπήρχαν ε, οι διοικητές των τραπεζών όπως και ο κύριος Μπαρνιέ και ε, ο κύριος Τρισέ. Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι προτάσεις για την νέα εποπτική αρχιτεκτονική και ε, συζητήθηκε επίσης και το μέλλον για την νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα. Επίσης ο κύριος Μπαρνιέ αναφέρει αναφέρθηκε στις ε, πρόσφατες ε, ε, συζητήσεις και στις επιπτώσεις. Εκτός αυτού, στην εφαρμογή στην Αμερική της νέας νομοθεσίας για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Επίσης αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει και μία ακρόαση για τις κρατικές βοήθειες και τους σχετικούς κανόνες που έχουν υιοθετηθεί μετά από την ε, οικονομική χρήση. Αύριο με 3 ε, με 6 το απόγευμα θα έχουμε μία δημόσια ακρόαση με τους κυρίους Μπανιέ και Αλμούνια και με τους ε, εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ε, σχετικά με την εφαρμογή ε, των κανόνων της κρατικής ενισχύσεως που εφαρμόζονται κατόπιν της οικονομικής κρίσης. Εάν λοιπόν έχουμε καταλήξει με αυτά τα θέματα, προχωράμε στο σημείο 3 της ημερησίας διατάξεως όπου έχουμε ε, μία έκθεση ΑΕΠ και πέρα από αυτό η μέτρηση της πρόοδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο για την οποία ε, ο εισηγητής είναι ο κύριος Νικόλαος Χουντής. Και έχει το λόγο. Συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος, όπως σύντομο είναι και το κείμενο της γνωμοδότησης και είναι σύντομο διότι σε αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εισαγωγή και άλλων δικτών μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο του ΑΕΠ ή εμπλουτισμού αυτού του δίκτυ, φαντάζομαι ότι όλοι θεωρούν ότι είναι ένα όριμο πρόβλημα που πρέπει να συζητηθεί. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε, το ΑΕΠ είναι το πιο διαδεδομένο στοιχείο και στατιστικό μέτρο για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Μετράει την προστιθέμενη αξία όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων Ωστόσο, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη που καταγράφεται στη γνωμοδότηση, η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί ένα μονοδιάστατο φαινόμενο. Δηλαδή μια διαδικασία την οποία να αυξάνει Η οικονομική ανάπτυξη έχει κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες δίκτυο. η οικονομικη αναπτυξη εχει κοινωνικες και περιβαλλοντικες πτυχέ, οι οποίε οφειλουμε οφειλει η επιτροπη να τις λαμβάνει υπόψη όταν καταγράφει το στατιστικό δυναμικό, όταν καταγράφει το ΑΕΠ. Δυστυχώ μέχρι τα τώρα κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα όπω η φτώχεια, η ανεργία, οι ανισότητε, η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του φυσικού πλούτου ε, που έχουν ενταχθεί κατά την έννοια του διαλόγου για τι οικονομικέ πολιτικέ δεν έχουν ενταχθεί, δεν περιλαμβάνονται στο δίκτυ και η πρόθεση που βάζει η ανακοίνωση τη Επιτροπή είναι ότι να βρεθεί τρόπο να ενταχθούν αυτέ οι δραστηριότητε. Αυτό σημαίνει, θα έλεγε κανεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση τότε στο ΑΕΠ θα έχουμε αυξομοίωση του ΑΕΠ αν έχουμε προβλήματα στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πλευρές. Ε, ε, επομένως, η γνωμοδότηση χαρακτηρίζει θετική αυτή την προσπάθεια που κάνει η Επιτροπή. Θετικό το γεγονός ότι προθεί πέντε δράσεις, δεν τις αναφέρω, είναι γνωστές, προκειμένου να βελτιώσει τη μέτρηση προόδου. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι πέρα από το ότι πρέπει να βελτιωθεί με περιβαλλοντικούς, με κοινωνικούς δείχτες η μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης, είναι φανερό ότι το πιο βασικό είναι ότι πρέπει στην διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι πτυχές. Δυστυχώς, το σημερινό κυρίαρχο καπιταλιστικό μοντέλο λαμβάνει υπόψη του κυρίως το κέρδος και αυτό καταγράφεται στο ΑΕΠ, ενώ τα άλλα ζητήματα είναι σε δεύτερη προτεραιότητα. Επομένως, Βεβαίως, θετική προσπάθεια να ενσωματωθούν οι πλευρές αυτές στη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά πιο σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές που να τα λαμβάνουν υπόψη από την αρχή και στο σχεδιασμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Um, the next Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Εσέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Χουντή. Συμφωνώ μαζί του ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική για να υπάρξει ε, ένα σοβαρός και ε, αποδοτικός ε, διάλογος επί του θέματος. Πιστεύω ότι σαν συγητής πρέπει να ζητήσει οι δημόσιες και οι ιδιωτικές αρχές να λάβουν υπόψη τους ε, τις κοινωνικές πτυχές των πράξεων αυτών και των ενεργειών αυτών. Εγώ έχω αμφιβολίες όσο για την δυνατότητα να υπάρξει ένας ενιαίος δείκτης. Εγώ θα μιλούσα μάλλον για, μία, ε, για ένα σύνολο ε, δείκτων και να βασιστούν και σε σωστές στατιστικές. Διότι τι σημασία έχει να έχουμε περίπλοκους δείκτες ε, εάν βασίζονται σε ασαφείς στατιστικές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε ε, καλά στατιστικά στοιχεία για να βασίσουμε τους δείκτες μας σε αυτά. Ε, και μετά νομίζω ότι ο εισηγητής απλώς απλοποιεί κάπως το οικονομικό μας σύστημα. Δηλαδή λέμε ότι απευθυνόμαστε ε, πρωταρχικά στην αύξηση και μεγιστοποίηση του κέρδους. Ενώ στην ε, Σκανδιναβία έχουμε ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο αποβλέπει στην ευημερία των πολιτών. Αντιλαμβάνομαι την άποψή σας αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικά τονισμένη η μεγιστοποίηση του κέρδους. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχουμε μία επικοδομητική συζήτηση για αυτή την γνωμοδότηση και χαίρομαι που συμμετέχω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έπινγκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ΑΕΠ είναι ένας βασικός δείκτης για την οικονομία και την οικονομική ζωή, διότι αποδεικνύει την απόδοση μίας χώρας, την παραγωγικότητά της και τους καθαρούς πραγματικούς μισθούς. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί πρέπει να μειώσουμε αυτό το πολύ καλό φαινόμενο γιατί θα καταλύσουμε σε ε, μαγικές οικονομικές ε, ε, μελέτες και η ερώτησή μου είναι πόσο όλα, όλες αυτές οι καλές προθέσεις θα ενσωματωθούν στις στατιστικές. Μιλάμε για τις κλιματολογικές αλλαγές. Αν υπάρχουν κλιματολογικές αλλαγές, πώς επηρεάζουν τις ε, χώρες, ε, πόσο, ε, πώς θα λάβουμε υπόψη μας την κοινωνική, την κοινωνική κάλυψη, διότι στη Γαλλία βλέπουμε ότι είναι δυσαρεστημένοι οι πολίτες με το σύστημα που έχουμε. Εάν λοιπόν προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα λέει ένα και ένα ίσον τρία γιατί φαίνεται πιο ωραίο θα το υιοθετήσουμε, διότι το μόνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα σας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Οπότε ε, δεν πρέπει να έχουμε μία ιδεατή οικονομία η οποία δεν θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή ε, υπηρεσία. Όλα αυτά προέρχονται από ε, ένα ωραιοποιημένο χώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος εξειδανικεύεται ακόμη περισσότερο στο Κοινοβούλιο και καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ένα παραμυθάκι που δεν πείθει ούτε τους πολιτικούς ούτε βεβαίως τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί πράγματι μιλάνε για παραμύθια. Όταν μιλάει κανείς για το ΑΕΠ δεν είναι ικανοποιημένος και υποστηρίζουν ότι ε, θα πρέπει να υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο η κατάσταση των οικονομικών κάθε χώρας. Βέβαια το ΑΕΠ το χρησιμοποιούμε εδώ και 50-60 χρόνια. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και μάλιστα έχουμε δώσει και βραβείο Νόμπελ σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι κάποιοι δείκτες θα πρέπει να προσπαθούν να μετρούν και την ευτυχία και όχι μόνο κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει αυστηρά οικονομικά στοιχεία και αριθμούς. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την έκθεση Στίγκλιτς σαν παράδειγμα Προτείνεται και εκεί να προσμετρηθεί με διαφορετικό τρόπο η ποιότητα της ζωής και να συμπεριληφθεί και η αηφορία, η αηφόρος ανάπτυξη στον υπολογισμό για την μέτρηση της, αηγο, της ευημερίας μιας χώρας. Αυτό είναι κάτι που θα συμπληρώσει τα στοιχεία τα οποία μας δίνει το ΑΕΠ. Έχουμε ανάγκη από οι οποίοι να αντικατοπτρίζουν κυρίως την πραγματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Για να τον πετύχουμε απαιτείται ένα συντονισμένος τρόπος προσμέτρησης των χαρακτηριστικών της οικονομίας και της κάθε χώρας και να κρίνουμε και τις κοινωνικές καταστάσεις και τις κοινωνικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Οι συζητήσεις αυτές με κάνουν ευτυχή. Εσείς που μιλήσατε προηγουμένως πιστεύετε ότι και ο εισηγητής, ότι και διάφοροι άλλοι οικονομολόγοι στην ουσία προτείνουν κάποιες οικονομικές πρακτικές που μοιάζουν σε βουντού και είναι μάλλον ανορθόδοξες. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ισχύσει για όλους, όχι μόνο για τον εισηγητή. Έχουν πράγματι εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες οι απόψεις που έχουμε για την καταμέτρηση της ευημερία μιας χώρας. Παράδειγμα, όσο περισσότερους, όσα περισσότερα περιπτώσεις καρκίνου σαν παράδειγμα έχει κανείς, όσο μεγαλύτερη καταστροφή υπάρχει, όσο περισσότερα τάνκερ σαν παράδειγμα να βαγούν και δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα, τότε τα χρήματα τα οποία δίδονται για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων καρκινοπαθών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των περιβαλλοντικών καταστροφών, χρησιμοποιούνται για να προσμετρηθεί προς τα πάνω η ευημερία μιας χώρας. Αυτό λοιπόν είναι voodoo economics, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει κάτι περίεργο, λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να βρούμε και άλλους δείκτες. Δεν λέει να απορρίψουμε τους προηγούμενους δείκτες. Εγώ δεν μπορώ να οδηγώ το αυτοκίνητό μου μόνο κοιτώντα τον δείκτη τον χιλιομετρικό. Δεν, δεν, δεν, δεν είναι δυνατόν. Σαν παράδειγμα εγώ χρησιμοποιώ και τον δείκτη κατανάλωσης καυσίμου που δεν είχε ο πατέρας μου όταν οδηγούσε αυτοκίνητο και φροντίζω καλύτερα την κατανάλωσή μου και είμαι πιο έξυπνος οδηγός. Φυσικά ένας οδηγός δεν μπορεί να βλέπει δέκα δείκτες ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε δεκάδες δείκτες γιατί δεν είμαστε και ουσιαστικά ικανοί να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα στοιχεία για να καταλήξουμε σε πολιτικές γραμμές. Πρέπει λοιπόν εμείς να φτιάξουμε ένα πίνακα με κάποιους λίγους βασικούς όμως δείκτες για να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Στη δουλειά στην οποία ασχολήθηκα πριν έρθω εδώ λένε ότι ό,τι μετρήσεις αυτό θα έχει στη διάθεσή σου. Λοιπόν, ό,τι δεν μετρήσεις προφανώς ε, δεν θα σε βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Το να προσμετρήσουμε σαν παράδειγμα τις κλιματολογικές αλλαγές ε, δεν είναι και κάτι το οποίο θα μας δώσει πολλά στοιχεία τώρα. Δεν μιλάω τώρα για την Ινδία, για την Κίνα, όπου πράγματι η αύξηση του ΑΕΠ βοηθάει τον κόσμο να ξεφύγει από την φτώχεια. Στις αναδυόμενες ε, οικονομίες υπάρχει ο συσχετισμός ανάμεσα στην αύξηση ε, του ΑΕΠ από τη μία και στην έξοδο των πληθυσμών από τη φτώχεια από την άλλη στις υπόλοιπες περιοχές βλέπει κανείς να υπάρχει μια αποσύνδεση ανάμεσα στην αύξηση του ΑΕΠ και στη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης. Μια αποσύνδεση της αύξησης του ΑΕΠ από τη μία και της ανόδου της φτώχειας από την άλλη. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για την σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη, την οικονομική από τη μία και την κατανάλωση των πρώτων, των πρώτων υλών από την άλλη. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε παρά να δούμε και άλλα πράγματα και άλλους δείκτες όπως αυτό το παράδειγμα που σας έδωσα για την κατανάλωση καυσίμων στο αυτοκίνητό μου. Λοιπόν, όχι πολλούς δείκτες, λίγους δείκτες, αλλά πρέπει φυσικά κάποιος να κάνει αυτές τις μετρήσεις και αν θέλουμε να έχουμε ισχυρά δεδομένα είναι σαφές ότι θα πρέπει η Eurostat να είναι το αποκλειστικό σώμα το οποίο να συλλέγει τα δεδομένα αυτά. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε 12 ιδρύματα που να κάνουν αυτό το πράγμα. Το Eurostat αν του δίνουμε καλά στοιχεία προφανώς θα κάνει καλή δουλειά. Βέβαια του έχουμε δώσει και λάθος στοιχεία και δεν έχει κάνει καλή δουλειά αλλά δεν είναι εκεί η ευθύνη. Λοιπόν είναι η πιο σοβαρή στατιστική υπηρεσία και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει πρωτοποριακά θα πρέπει να ζητήσουμε από την Eurostat να αρχίσει να συλλέγει δεδομένα για τις ανισότητες της κοινοτικέ. Αυτό μετράται. Σαν παράδειγμα κατανάλωση πόρων και αποτελεσματικότητα στην κατανάλωση πόρων και πρώτων υλών. Τέτοιου είδους δείκτες είναι απαραίτητοι, ακόμα και πέραν από αυτούς τους δείκτες. Εμείς ασχολούμεθα, ας πούμε, με την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Έχουμε και τον εισηγητή εδώ γνωρίζουμε ότι σαν τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα έχουμε και το λεγόμενο dashboard των πίνακα στόχων που ε, θα δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά Στη συνάντηση που είχαμε με την Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2011, σύντομα δηλαδή, να συμπεριλάβει και κάποια στοιχεία κοινωνικού τύπου, κοινωνικές ανισότητες, περιβαλλοντικού τύπου, περιβαλλοντικές μετρήσεις στην έκθεσή του. Αυτό δείχνει ότι ναι μεν δεν θα έχουμε κάτι το πλήρες, αλλά ήδη από τώρα μπορούμε να έχουμε κάποια πρώτα αρχικά στοιχεία. Δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ήδη σαν σκληρά στατιστικά δεδομένα για να προσμετρήσουμε ε, την οικονομική κατάσταση μιας χώρας, αλλά σίγουρα θα αρχίσουμε να συλλέγουμε τέτοια στοιχεία για να εκτιμήσουμε κάπως τα πράγματα διαφορετικά. Πρέπει να δει θάρρος γιατί είπαμε αυτό το οποίο θα πάρουμε είναι αυτό το οποίο θα θελήσουμε να μετρήσουμε. Νομίζω ότι είναι περίεργο μια τέτοια σύσταση να προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και να πηγαίνει στην συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι το θέμα της καταμέτρησης όλων αυτών των δικτών είναι δική μας αρμοδιότητα και όχι της Επιτροπής Περιβάλλοντος, σαν παράδειγμα γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύστημα έτσι ώστε τα στοιχεία τα οποία θα προέλθουν από τη συλλογή αυτή που θα γίνει να μην ληφθούν και πολύ σοβαρά υπόψη στην κατάρτιση των πινάκων με τις επιδόσεις της κάθε χώρας. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Καταλαβαίνω τα σχόλια της ΕΣΑΙΑΣ ότι δεν πρέπει να υπεραπλουστεύουμε σχετικά με το υπερβολικά κέρδη κτλ. Όταν έφυγε από την επιχείρηση στην οποία δούλευα εδώ και ένα χρόνο, το μόνο πράγμα το οποίο μετρούσαμε ήταν το κέρδος. Α μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό ισχύει γενικά στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι πολιτικοί έχουν μόνο αυτό στο νου τους, αλλά είναι σαφές ότι η οικονομία της αγοράς όσο τρέχει έτσι ανεξέλεγκτη το μοναδικό πράγμα το οποίο κυνηγάνε είναι ένα, ο μοναδικός δείκτης τον οποίο κυνηγάνε είναι ένας, όχι μεσοπρόθεσμα ή, βραχυπρό, ή μακροπρόθεσμα κέρδη, αλλά βράχυπρόθεσμα τα μέγιστα κέρδη. Εμείς δεν θέλουμε να μειώσουμε τα κέρδη αυτά. Θέλουμε όμως να το συνδυάσουμε και με κάποιες άλλες μετρήσεις οι οποίες για μας έχουν σημασία. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μετά από τον Φίλιπ Λάμπερτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω κάτι από τον κόσμο τον πραγματικό και όχι από τον κλειστό κόσμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούσατε προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Λάμπερτ γιατί και αυτός έρχεται από τον έξω κόσμο σε εισαγωγικά και έχει και κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με μένα. Ένα από αυτά είναι ότι ο Λάμπερτ προέρχεται από ένα κόμμα το οποίο σε διάφορες περιοχές ε, σημαντικών χωρών έρχεται κοντά στην εξουσία πλησιάζει την εξουσία. Οπότε αυτά που λέει ο Λάμπερτ θα μπορούσε να τα πει και ένα πρωθυπουργό κάποτε και ένα πρόεδρο δημοκρατία κάποτε. Λοιπόν έχουν σημασία αυτά που λέει. Αν λειτουργήσω με την ίδια διαδικασία της, α, της απόσυρσης και αντιγραφής του copy-paste, εν πάση περιπτώσει των υπολογιστών, τότε αυτά που ακούσαμε θα μπορούσε να τα πει και κάποιος εκπρόσωπος του Πρασίνου κόμματος. Δεν θέλω τώρα να πω ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε το copy-paste του Λάμπερτς και ότι μαζί με τους πρασίνους θα πετύχουμε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για όλους. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Αυτό που θα έπρεπε να πω είναι ότι θα περίμενα κάπως περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία στη γνωμοδότηση αυτή. Παρ' όλα αυτά μπορώ να παρακολουθήσω τη γνωμοδότηση, και συνοπτικά να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπα την προηγούμενη εβδομάδα όταν παρουσίασα τη γνωμοδότησή μου για την οικονομική διακυβέρνηση, τη γενική εικόνα πάνω στην οποία θέλουμε να δουλέψουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι τότε υπήρχαν μόνο δύο-τρεις συνάδελφοι στην αίθουσα ε, και τώρα που είναι πιο βασικό το θέμα ε, μπορούμε να προσελκύσουμε και πιο νέους στο θέμα αυτό το οποίο είναι ε, σημαντικό και να επιτύχουμε να εφαρμόσουμε την αρχή ότι data can be sexy. Βέβαια βλέπουμε ότι υπήρξαν κρίσεις στην Ελλάδα και σε άλλες άλλες και υπάρχει επιρροή στην ευημερία των πολιτών και όταν φτάνετε εις ε, το Βέλγιο βλέπετε ότι παντού υπάρχουν πινακίδες που σας υποκινούν να προχωρήσετε στην επόμενη, στο επόμενο επίπεδο αναπτύξεως, πράγμα το οποίο θα έπρεπε να ισχύσει παντού. Βέβαια θα έπρεπε ε, να υπάρχουν στατιστικές της ε, ευρωπαϊκής αηφορίας κατά τρόπον ώστε να δούμε ποια είναι είναι τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της ε, ευρωπαϊκής ε, ε, πολιτικής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρότυπα διότι ε, εκτός από τα στιγμιαία πρότυπα ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τύπους που περιλαμβάνουν ε, διάφορους λογαριασμούς τις πρώτες ύλες, το νερό, την ενέργεια δηλαδή όλα αυτά δεν προέρχονται από μία αρχική σκέψη των πρασίνων και εγώ είχα εμπλακεί στο παρελθόν ε, σε μία ομάδα εργασίας του Eurostat και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Eurostat, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία και να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να πούμε ναι αντιλαμβανόμαστε ότι οι δείκτες που έχουμε για την ευημερία δεν επαρκούν και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και νέους και να υπάρχουν ε, να υπάρξουν και νέα στοιχεία ανταγωνιστικά αλλά αυτά κοστίζουν χρήματα. Χρειαζόμαστε έμπειρους και οι πράσινοι ε, στο σημείο αυτό και η ε, θέση που εγώ και πολλοί ψηφοφόροι εκπροσωπούν ε, δεν συνάδουν. Μπορούμε όμως να χρηματοδοτήσουμε την προσπάθεια αυτή εάν ασχοληθούμε με την ε, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή μετά από τόσες διευρύνσεις προς τόσα κράτη δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ε, επαρκής ε, επαρκής ε, έμπειρη γνώμη που θα μπορούσε με κάποια μετάθεση να χρησιμοποιηθεί ε, πιο αποδοτικά. Δηλαδή πρέπει να μειώσουμε την και γραφειοκρατία, πρέπει να έχουμε ένα διευρυμένο στατιστικό δίκτυο στην Ευρώπη κατά τρόπον ώστε να παρακολουθούμε την ανάπτυξη υπορεαλιστικούς όρους και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε μια, προσωπικη σε μια μια προοπτική η οποία δεν θα αναφέρεται μόνο στην πρόοδο όπως την εννοούμε τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Μαν, παρακαλώ να είστε σύντομος για να μπορέσουμε να συνοψίσουμε. Ναι κύριε Πρόεδρε, θα είμαι ε, σύντομος, δεν θα πλατιάσω σαν τον προλαλήσαντα, παρόλο που ε, βλέπω ότι οι πράσινοι κινούνται στη μέση και το είδα αυτό και στην ε, ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπου υπάρχουν δημοκρατικές αρχές, τις δέχομαι και ίσως αυτό οφείλει λέτε ότι όλοι θέλουν να καλύψουν το αστικό ε, ε, κέντρο, δηλαδή το, τους ψηφοφόρους οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο και απέχουν από τα άκρα. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Μάρτιν είναι σωστό υπάρχουν πάντοτε οι σκέψεις να λέμε ότι ε, η Ευρώπη επεμβαίνει πάρα πολύ πολύ ε, ενώ χρειαζόμαστε περισσότερα στατιστικά στοιχεία. Άρα πρέπει να νομιμοποιηθεί και η Eurostat για να μπορεί να συλλέγει, να αναλύει στοιχεία τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε όλοι. Άρα δεν χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη αλλά περισσότερη Ευρώπη θα είναι μια πολύ θετική στάση την οποία πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Και αυτό ισχύει και σε άλλα θέματα, στα θέματα του περιβάλλοντος, της αηφορίας και όλα αυτά είναι κέρδος διότι ε, αν μπορέσουμε να τονίσουμε τις διαφορές και να ενισχύσουμε το κέντρο πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερες δυνατότητες. Πιστεύω ότι η γνωμοδότησή σας είναι καλή η οποία τονίζει τα βασικά θέματα και θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε το κέντρο, τον πυρήνα ε, και την περιφέρεια της Ευρώπης μαζί με την έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, ε, βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι κοιτάζει κανείς τα θέματα από διαφορετικές σκοπιές αλλά η συζήτηση αυτή ε, γίνεται πολύ καιρό τώρα και με ακαδημαϊκούς και με πανεπιστημιακούς λέμε ότι ο τρόπος αξιολογήσεως του ΑΕΠ δεν είναι τέλειος και ξέρω ότι έχουμε προσπαθήσει να βρούμε δείκτες αηφορίας και να καθορίσουμε ε, διάφορες μοφές εργασίας και ε, αξιολόγησης των διαφόρων μορφών εργασίας. Λοιπόν, ε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε επικαλύψεις αν αυτά συζητούνται σε διάφορα άλλα σημεία εκτός του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, Eurostat να συνεργάζεται με τον ΩΣΑ διότι ακόμη και ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχει δείκτες οι οποίοι είναι γενικώ αποδεκτοί οπότε να ας στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και όταν θα έχουμε αρκετές γνώσεις που να αποδεικνύουν ε, ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε προβλήματα θα μπορέσουμε ίσως να μετρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το οποίο επιζητούμε. Ζητώ λοιπόν τώρα από τον κύριο Χουντή να παρουσιάσει τα συμπεράσματα της συζητήσεως που είχαμε μέχρι τώρα και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που έγιναν νομίζω επιβεβαιώθηκε ότι αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο έχει βάση. Η γνωμοδότηση προφανώς είναι σύντομη, ενδεχομένως και από τους περιορισμούς που τίθενται γραμματιακά μέσα σε μισή σελίδα, μια σελίδα, να γράψεις ποια είναι η γνώμη σου σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής. Η συζήτηση όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που ζητάει η γνωμοδότηση να πούμε είναι θετικό αυτό, να ξεκινήσει, να προχωρήσουμε. Ε, η δεύτερη μου παρατήρηση. Δεν ε, υιοθετώ την άποψη που ακούστηκε ότι καλό είναι το ΑΕΠ, α μείνουμε σε αυτά, μην μπλέκουμε με πολλού δείχτε, μπορεί να πάμε σε ένα χάο που δεν θα μπορούμε να βρούμε άκρη. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η τυπολογία, η τύπη στην οικονομική επιστήμη, σε μια προσπάθεια να μιμηθεί η οικονομική επιστήμη άλλε επιστήμε όπω τη φυσική και τα μαθηματικά, δεν απηχούν την πραγματικότητα. Τι πάει να πει δηλαδή έχουμε μείνει στο ΑΕΠ με το γνωστό τύπο ιδιωτική κατανάλωση και ούτω καθεξής. Και αυτό μπορεί να μετρήσει ένα ζωντανό πράγμα όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη και να περιφρουρήσουμε και να πούμε μείναμε εκεί. Δεύτερη, εμείς πολλές φορές στην Ελλάδα και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα λέμε πολλές φορές οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Δηλαδή η άνοδος του ΑΕΠ σε μια χώρα δεν σημαίνει πως έχει ασφαλίσει αντίστοιχη ευημερία για το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών δεν υποτιμώ τη μέτρηση του ΑΕΠ έτσι όπως γίνεται μέχρι τώρα. Πρέπει κάτι να μετριέται για να μπορείς να χαράξεις, να έχεις κάποιους στατιστικούς δείξεις, να χαράξεις την πορεία από εδώ και πέρα. Αλλά όμως η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι ότι σήμερα στοιχεία που συγκροτούν την ευημερία των πολιτών, που συγκροτούν την προστασία του περιβάλλοντος που έχει οικονομικές διαστάσεις, δεν μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη στην σχεδιασμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Επομένως, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια προσπάθεια στατιστικής μελέτης και στατιστικών δεδομένων. Αυτό λέει η γνωμοδότηση, έγιναν αρκετές παρατηρήσεις και η τρίτη τελευταία παρατήρηση καταλαβαίνω ότι και σε κάποιον που το αποδέχεται αυτό, λέει εντάξει να βάλουμε και τις κοινωνικές και τις παρεμβαλλοντικές πτυχές, ενδεχομένως βλέπει μπροστά δυσκολίες με ποιε τεχνικές θα μπορέσεις να μετρήσεις αυτές τις πτυχές, πτυχές που καλό θες να, να μπει εκεί. Από ό,τι είδα και από την ανακοίνωση και από ό,τι έχω διαβάσει, υπάρχουν μια τεχνογνωσία που αναπτύσσεται που μπορεί να μα δώσει τη δυνατότητα να πάμε σε πιο δείκτε, όχι πολλού όπω είπαν αρκετοί συνάδελφοι, αλλά εν πάση περιπτώσει να καταγράφουν αυτέ τι πτυχέ για τι οποίε όλοι νομίζω συμφωνούμε, συγκροτούν εν τέλει αυτό που θα λέγαμε οικονομική ε, ανάπτυξη. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Ε, Uh, Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 12 Οκτωβρίου. Εξέταση των τροπολογιών ε, θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 26 Οκτωβρίου. Στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος μεταξύ 29 Οκτωβρίου, ε, Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου και θα ε, ψηφιστεί στη, στο, στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου 2011. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2009. Ο κύριος Μπάλτς δεν είναι εδώ. Ίσως ο κύριος Γκοζές να θέλει να πάρει το λόγο. Président, effectivement, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάλτς μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόμασών του γιατί είναι σε αποστολή ε, με το Ίδρυμα Κόντραντα Ντενάουερ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάσατε την έκθεσή του. Ο κύριος Πάλτς μου ζήτησε, επειδή δυστυχώς δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα, να ευχαριστήσει όλους όσους επέβαλαν τροπολογίες και μου είπε επίσης ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό ε, των διαφόρων τροπολογίων. Αυτό έχει φανεί και από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Δεν υπάρχει σοβαρή διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ε, μπορεί να αξιολογήσει κανείς την έκθεση της ΕΚΤ. Κατά την άποψή του είναι αποδεκτές οι τροπολογίες και για κάποιες από αυτές που θα μπορούσε να γίνει συζήτηση προτείνει να συναντηθεί με τους υποβάλλοντες τις τροπολογίες για να βρεθεί ένας ε, συμβιβασμός. Είναι σημαντικό για να έχει αντίκτυπο η έκθεση αυτή να είναι αντικείμενο μεγάλης συνένεσης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό ζητά από τους χειόδους εισηγητές ε, να μην διστάσουν να έρθουν σε επαφή μαζί του για να ε, συζητηθεί το, τελευταίο, το τελικό κείμενο. Κατά τη διάρκεια του Στρασβούργου ζητά να ε, καταλήξει σε συμβιβασμό για να μπορέσουμε να, μπορέσουμε να ψηφίσουμε το θέμα στις 26 Οκτωβρίου. Αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες που μου ζήτησε να σα μεταβιβάσω. Θα σημειώσω βεβαίω τα σχόλια των συναδέλφων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. αν Uh, Υπάρχουν uh, σκιώδεις uh, εισηγητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Κούτας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλς γιατί επέδειξε ευρύτητα πνεύματος. Συζήτησα κάποιε τροπολογίε μαζί του σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, που κατά τη γνώμη μα είναι περιορισμένο εργαλείο για την ε, επίλυση του ζητήματο των οικονομικών ανισοτήτων. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη ε, φιλόδοξη μεταρρύθμιση ε, του Συμφώνου που θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυση της συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Επίσης θα ήθελα να πω για το χρέος ε, της Ευρωζώνης ε, που ήταν προβληματικό κατά τη διάρκεια ε, της κρίσης. Φάνηκε δηλαδή το πρόβλημα και γι' αυτό θα θέλαμε να εξετάσουμε το θέμα των οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Θα ήθελα να υποστηρίξω επίσης αυτό που είπε ο κύριος Σικλούνα για το πρόβλημα των περικοπών των δημοσιονομικών τη στιγμή που δεν έχει ανακάμψει ακόμη η ευρωπαϊκή οικονομία. Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο σας. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις και αυτός είναι ο λόγος ε, που ε, οι τράπεζες είναι λιγότερο πρόθυμες να δανείσουν και όχι ο λόγος που αναφέρεται στην τροπολογία 66. η κρίση έχει ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό βέβαια επηρεάζει την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Λάμπερτ ότι η ΕΚΤ πρέπει να λάβει υπόψη τις διαφορετικέ διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των οικονομιών που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ε, στρατηγική ε, εξόδου από την κρίση, κάτι το οποίο αναφέρεται στην τροπολογία 76. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε κούτα. Η Σοφή Νετβέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Κοίταξα λίγο τις τροπολογίες και μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλές από τις τροπολογίες αυτές. Υπάρχουν όμως ορισμένες τροπολογίες οι οποίες τι λέγουν. Λέγουν ότι η αποτυχία στην προσπάθεια μεθαρρύθμισης μπορεί να αντισταθμιστεί με την ύπαρξη υψηλότερων χρεών και ελλημάτων. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό αυτό. Είμαστε υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχία και υπέρ της λειτουργίας του Συμφώνου Ανάπτυξης. Αυτή είναι η στάση της πολιτικής μας ομάδας όταν κρίνουμε μεμονωμένα α, τις τροπολογίες αυτές. Φυσικά θα υποστηρίξουμε θετικά τις πράσινες τροπολογίες, κάποιες από τις δικές σας, αλλά όχι τις τροπολογίες Κλούιτε. Νομίζω ότι έχω καλύψει τις περισσότερες από τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Μάννα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αν ήταν εδώ ο συνάδελφος θα είχα κάνει ερωτήσεις αλλά θα τους διαβιβάσει ίσως ο Ζων Πολ. Όσον αφορά την τροπολογία 51 ελέγχθη ότι η ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζά θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαφάνεια. Πράγμα όμως το οποίο γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο έχουμε συνεδριάσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο κύριος ε, Τρίσε έχει συμμετάσχει επανειλημμένου στις συνεδριάσεις μας άρα πιστεύω ότι πρόβλημα υπάρχει περισσότερο με τροπολογία 52 γιατί ζητάμε να δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων διότι αν ε, τα μελετήσουμε και δούμε τι διαφορές υπάρχουν θα δείτε ότι όντως μπορεί να υπάρξει μία ενιαία συμφωνία των, των διαφόρων απόψεων και εάν κοινοποιόντουσαν τα πρακτικά θα μπορούσε να διεπιστώσει και το κοινό ότι υπάρχει μία σύμπνοια αλλά ναι μεν υπάρχει ανεξαρτησία, ναι υπάρχει διαφάνεια αλλά ε, ε, πιστεύω ότι ε, τα πρακτικά δεν με βρίσκουν τόσο σύμφωνο στο να δημοσιεύονται. Ε, μετά, ε, λέγεται ότι το ευρώ είναι ισχυρό. Βέβαια δεν είναι καλό, διότι είναι κακό για τις εξαγωγικές μας βιομηχανίες. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και ο αντίλογος, αν είναι πιο αδύναμο. Εάν το ευρώ είναι σταθερό, τότε ε, υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους πολίτες μας, οι οποίοι είχαν πει ότι εάν έχετε ένα κοινό νόμισμα, ποτέ δεν θα είναι ισχυρό, ποτέ δεν θα είναι σταθερό, άρα το, το ζητούμενο δεν είναι να είναι χαμηλή ισοτιμία για να μπορούμε να εξάγουμε, αλλά να υπάρχει περισσότερη ισορροπία και να είναι σταθερό το νόμισμα. Οπότε την ε, τέταρτη τροπολογία δεν συμφωνώ, αλλά κατά τα άλλα όσον αφορά τις περισσότερες θέσεις πρέπει να σας πω ότι δεν, ε, δεν έχω αντίρρηση στα υπόλοιπα θέματα. Θα συστήσω άλλωστε και στην ε, πολιτική μου ομάδα να συνενέσει και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε ένα συμβιβασμό. Ζων Πολ, θα σου μιλήσω γαλλικά. Πρώτα απ' όλα, Καταρχήν είχαμε μία συζήτηση με τον εισηγητή τον κύριο Μπάλτς και είδαμε ότι συγκλίνουμε σε πολλά σημεία. Εφιστώ την προσοχή λοιπόν σε δύο θέματα. Καταρχήν ο εισηγητής έχει πρόβλημα με ορισμένες τροπολογίες τις οποίες έχουμε υποβάλει ε, ιδίω για τη διαφάνεια. Άκουσα τις, ε, τα σχόλια του κυρίου Μαν για την ε, δημοσίευση των πρακτικών αλλά ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποίησε τα τελευταία χρόνια άτυπες ε, μεθόδους και πήρε άτυπα μέτρα ε, ξέρετε ότι όσοι ε, όσες εταιρείες τράπεζες δηλαδή χρηματοδοτήθηκαν εποφελήθηκαν πράγμα το οποίο όμως δεν ίσχυει για όλους Οπότε αναρωτιόμαστε ε, για το αποτέλεσμα των ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, στην, στον τομέα της, ε, του ανταγωνισμού, του ισοσχελισμένου ανταγωνισμού. Μήπως λοιπόν στήριξε τράπεζες οι οποίες είχαν ε, κακή ε, συμπεριφορά. Άρα αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, να ξέρουμε ποια είναι η φύση των μέτρων, ποιος επωφελήθηκε και μία ανάλυση για να δούμε πώς επηρέασαν τον ανταγωνισμό. Και τέλος συμφωνώ με αυτό που είπε η Σοφή Δηλαδή, εμείς μιλάμε για τις αιτήσει εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι για την μακροοικονομική πολιτική στην Ευρώπη. Θα έχουμε, το είδαμε την έκθεση Φεγιό, θα το δούμε με τις έξι εκθέσεις για την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άρα πρέπει να αποφύγουμε τον πειρασμό να προσπαθούμε να βάζουμε τα πάντα σε, σε κάθε συζήτηση Άρα όταν μιλάμε για την ε, ανάλυση των ε, λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν πρέπει να αναμειγνύουμε άλλα θέματα και καλύτερα αυτά τα άλλα θέματα να μείνουν εκτός αυτής της εκθέσεως. Ευχαριστώ. Μία μικρή διευκρίνηση. Και εγώ όπως και οι συνάδελφοί μου θεωρούμε ότι είναι μια καλή έκθεση, έκθεση μπάζ. Οι τροπολογίες είναι χρήσιμες και ελπίζω να υπάρξει μια συμφωνία. Ένα ειδικό θέμα αφορά το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας. Όλοι συμφωνούμε ότι τα μέτρα της λιτότητας ή τα μέτρα εν πάση περιπτώσει φορολογικής και οικονομικής εδραίωσης είναι μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις οικονομίες να ανακάμψουν. Αν δεν είχαν ληφθεί η κατάσταση θα ήταν χειρότερη. Αλλά σε μια εποχή όπου η οικονομία είναι πραγματικά εύθραυστη, τέτοιου είδους μέτρα εξοικονόμησης ταυτόχρονα σε πάρα πολλές χώρες, απαιτεί τη σύνδρομή των κεντρικών τραπεζών. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μικρό περιθώριο γιατί τα επιτόκια είναι ιστορικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να διασφαλίσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει όπλα για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας τα οποία παίρνονται ομαδικά στις οικονομίες μας πλέον. Ο κύριος Γκοζές για να κλείσει τη συζήτηση. Θα ήθελα να πω στον καθένα από τους ομιλητές ότι πράγματι σημείωσα τις τροπολογίες που τους δημιουργούν κάποια προβλήματα και θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις τους στον κύριο Μπάλς. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε ο προηγούμενος συνάδελφος θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιες αρνητικές ε, συνήθειες που έχει η Επιτροπή Γυναικών του Κοινοβουλίου μας, η οποία θέλει συνέχεια να φτιάχνει εκθέσεις, οι οποίες ψηφίζονται μέσα σε πέντε λεπτά και σε πέντε λεπτά στην Ολομέλεια και που αφορούν το ίδιο θέμα και επικαλύπτουν η μία την άλλη. Γι' αυτό ακριβώς είχα κάνει την παρατήρηση που έκανα και στην ημερήσια διάταξη έχω την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε στις εκθέσεις αυτές θέματα τα οποία φύγουμε σε άλλες εκθέσεις και σε μελλοντικέ εκθέσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Επιμένω γι' αυτό γιατί είμαι μόνιμο θύμα στην Επιτροπή Γυναικών αυτή της απαράδεκης πρακτικής και προσπαθώ πάντα στην Ολομέλεια να επανορθώνω την κατάσταση, δεν το πετυχαίνω πάντα, μερικές φορές μόνο. Πρέπει αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να πάρει τον εαυτό της σοβαρά και να μην επαναλαμβάνει μονίμως τα ίδια πράγματα. Καλώς. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι η ψηφοφορία θα γίνει την 26η Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας και το Νοέμβριο πάντα θα έρθει και στην Ολομέλεια τη δεύτερη. Η συζήτηση ε, της 22ης Νοεμβρίου με τον κύριο Τρισέ είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσετε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι το σημείο 6. Είναι το κείμενο εργασίας για τις καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης. Α, για μια στιγμή υπάρχει κάτι, κάποιο θέμα εδώ. Συγγνώμη David, κάτι ξέχασα. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση για το κοινό σύστημα ΦΠΑ. Αφορά τη διάρκεια της υποχρέωσης σεβασμού ελαχίστου ποσοστού επιβολής. Ε, ο κύριος Κάζα είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε ότι από το 1993 οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να έχουν έναν ελάχιστο ε, φόρο προστιθέμενης αξίας ε, του 15%. Το 1993 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει μια εναρμονισμένη δομή ε, και πρότεινε ένα χαμηλότερο ε, ΦΠΑ με ένα κατώτατο όριο. Ε, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, λήψη πολιτικής συμφωνίας που είχε ως αποτέλεσμα την συμφωνία που ανέβαλε ουσιαστικά την εφαρμογή του συστήματος αυτού, εισήχθη το σύστημα που ισχύει σήμερα. Τέσσερις παρατάσεις πήρε η συμφωνία αυτή και θα, ολοκληρώ, θα, θα εκπνεύσει στο τέλος του τρέχοντος έτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί για ακόμη πέντε χρόνια. Το τρέχον σύστημα ε, είναι μεταβατικό, δεν ε, συνάδει για πολλούς λόγους με την εσωτερική αγορά και πρέπει να γίνει μια διαδικασία διαβούλευσης ε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον καλύτερο ε, τρόπο να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου είπε ότι θα υπάρξει και πράσινη βίβλος για αυτό το θέμα σύντομα ε, και ότι θα τη λάβουμε πολύ σύντομα. Εγώ βέβαια θα ήθελα να μην βιαστούμε πάρα πολύ η διαβούλευση να γίνει ε, με τρόπο ε, που να είναι έγκαιρος και αποτελεσματικός. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να συμμετέχει το συντομότερο δυνατόν. Ελπίζουμε οι επακόλουθες νομοθετικές προτάσεις ε, να συμπεριλάβουν ε, στις αποφάσεις ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το λέω αυτό εν ώψη της αναθεώρησης που θα γίνει το 2013. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και αναμένω εναγωνίως τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών προκειμένου να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαμπέρτς. Ευχαριστώ. Την τιμητική μου έχω σήμερα το απόγευμα. Για το ΦΠΑ. Η παράταση του τρέχοντος καθεστώ, καθεστώτος, ε, ελάχιστο φόρος δηλαδή 15%, σημαίνει δύο πράγματα. σε σχέση με το ΦΠΑ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι είναι πάντοτε ιδιαίτερη χαρά να ικανοποιούμε κάποια τμήματα του εκλογικού σώματος, ειδικότερα όταν έχουμε σοβαρές δημοσιονομικές περικοπές. Ε, πάντοτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε αγγελιοφόροι κακών νέων, το είδαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα ε, στους δρόμους με τις διαδηλώσεις των εργαζομένων. Ενδεχομένω να κάνουμε χάρες σε κάποιους κλάδους. Ξέρετε αυτό το ζήτημα της περικοπής του ΦΠΑ που είχαμε για τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία κατά τα τελευταία χρόνια για να ευχαριστήσουμε ουσιαστικά τον κλάδο αυτό, ενώ ζητούμε από άλλους να κάνουν ε, σοβαρή προσπάθεια, να κάνουν σοβαρές προσπάθειες. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ε, αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα. Δεύτερον, είναι το θέμα της ε, φοροδιαφυγής. Γνωρίζετε ότι εκτιμάται και εντάξει επειδή δεν ε, ε, αναφέρεται ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ γιατί πόσο μιλάμε, αλλά είναι περίπου 300 δισεκατομμύρια ε, κατ' έτο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να πει κανεί ότι θα πάμε στο μηδέν, ότι θα το μειώσουμε στο μηδέν, αλλά αν μπορούμε να πούμε ότι στα επόμενα 5-10 χρόνια θα έχουμε ε, μία στρατηγική για να το μειώσουμε, αυτό σημαίνει μεγαλύτερα έσοδα για τι κυβερνήσει και γνωρίζουμε ότι τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ για να χρηματοδοτήσουμε μελλοντικέ επενδύσει, ε, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση. Η φοροδιαφυγή ε, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να ε, προτρέχουμε σε σχέση με την ε, μεταρρύθμιση. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μια ευρεία πολιτική βάση για να ε, έχουμε ένα γνώμονα, τα κριτήρια επί των οποίων θα πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια αναθεώρηση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε πολιτική συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών οικογενειών, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε πάντοτε να περιμένουμε την Επιτροπή να μας υποβάλει προτάσεις. Θα μπορούσαμε κι εμείς πώς να το πω, να, ε, να επηρεάσουμε λίγο την υποβολή των προτάσεων αυτών από το να κάτσουμε να περιμένουμε να μας τις υποβάλουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εργασία του. Το θέμα ε, ε, αναφέρεται στην παράταση των προσωρινών μέτρων μέχρι ότου ισχύσει ο, ο κατώτατος γενικός συντελεστής ΦΠΑ. Και ε, δεν χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση οπότε η πρόταση ε, ουσιαστικά συνάδει με το στόχο που επιζητά για να μην υπάρχει επιπρόσθετο κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε για τις επιχειρήσεις ή για τους καταναλωτές. Όμως επειδή γενικώ συμφωνούμε με την πρόταση αυτή, θα ήθελα να σας πω ότι παρόλες τις βελτιώσεις, το κοινό σύστημα του ΦΠΑ υποφέρει από ελλείψεις και ε, δαπανηρό κόστος. Ε, και πρέπει να υπάρχει μια οικονομική επαναξιολόγηση γιατί η οικονομική ε, πραγματικότητα μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναξιολογήσει ε, τις νέες αυτές πραγματικότητες και να εκπονήσει μια νέα στρατηγική για αυτήν ε, την, την αξιολόγηση του ΦΠΑ χωρίς ε, όμως να παραβλέπουμε ότι χρειαζόμαστε γρήγορα ένα ε, τελεσίδικο πλαίσιο πριν ε, εκπνεύσει η ισχύ του προηγουμένου και η έκθεση Μόντι ούτως ή άλλως αποτελεί μια κατευθυντήριο γραμμή επί του θέματος. Ευχαριστώ κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Μπάις. Δηλαδή, τον κύριο Κάζα. Δηλαδή, ε, όταν πρωτοήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, προσπάθησαν να, να επαναφέρουν το σύστημα του ΦΠΑ και ε, απερίφθη πλήρως. Πιστεύω ότι το ΦΠΑ μέσω πολιτικών αποφάσεων δεν μπορεί να επηρεάσει τους πολίτες στην απόφασή τους το τι θα αγοράσουν ή τι θα κάνουν με τη ζωή τους αλλά ουσιαστικά είναι μία αποτυχία σε όλη την Ευρώπη διότι συμφωνώ ότι για το για τα εστιατόρια και τα λοιπά ήταν λαθασμένο και οι φίλοι μου στη χώρα μου το προτείνουν επίσης γιατί λένε ότι εφόσον είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό θα είναι καλό για μας αλλά δεν θα επωφεληθούν οι πολίτες και γι' αυτό καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στον Επίτροπο ότι θα πρέπει να κάνει αυτό το οποίο έκανε και ο κύριος Μπόλκερστάιν αλλά αν το πράξει θα πρέπει να τον στηρίξουμε διότι αυτό δεν έγινε την τελευταία φορά και το αποτέλεσμα του νέου προγράμματος ΦΠΑ μπολκενσταιν δεν ήταν λιγότερα ποσοστά ΦΠΑ αλλά μια από τα ίδια. Δηλαδή και πάλι τα κράτη μπορούσαν να επινοήσουν νέες μεθόδους για το ΦΠΑ οπότε συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κάζα. <coughs> Κύριε Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Κάζα, να συμφωνήσω με την γραμμή την οποία προτείνει, δηλαδή την δυνατότητα διεύρυνσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου του παρόντος καθεστώτου. Ξέρουμε ότι το καθεστώς αυτό δεν είναι καθόλου ιδανικό όταν ορίσαμε το κατώτερο ποσοστό ήδη το 1993 γνωρίζαμε ότι και επί τη βάση του φορολογικού ανταγωνισμού θα φτάναμε σε κάποια στιγμή στην γυρνίαση του ύψους ε, επιβολής. Δεν έγινε αυτό γιατί οι χώρες που είχαν υψηλή, ε, υψηλό επίπεδο επιβολής ΦΠΑ ε, το ανέβασαν ακόμα περισσότερο. Εγώ γνώρισα πάρα πολλούς επιτρόπους τα τελευταία χρόνια, Μπόλκενστάιν, Κόβατς και το μόνο που πρότειναν κάθε φορά ήταν να αυξάνεται το ποσοστό του ΦΠΑ και να μειώνονται οι δασμοί και τα τέλη, τα ειδικά στο ενόπνευμα, στον καπνό, στη βενζίνη κτλ. Δεν πρόσεξαν καθόλου τις διαφοροποιήσεις στο επίπεδο ε, ΦΠΑ. Βέβαια κάποιες από τις προτάσεις τους ευτυχώς δεν έγιναν δεκτές και κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα τώρα πλέον σε επίπεδο επιβολής φόρων. Και μάλιστα τελευταία μιλάμε όλο και περισσότερο για θέματα απατών και φοροαποφυγής και απαλλαγής γιατί δυστυχώς οι υπερβολικοί φόροι σκοτώνουν τον φόρο ουσιαστικά έτσι λέμε. Έχουμε κάνει και εκθέσεις γύρω από αυτό το θέμα. Δεν θέλω να ξεκινήσω εκ νέου τη συζήτηση, ιδιαίτερα για το μειωμένο ποσοστό επιβολής. Είχαμε τεράστιες συζητήσεις εδώ, ιδιαίτερα από την εποχή Μπόλκενστάινα. Μας είχε πει ότι όταν είχαμε αποφασίσει μειωμένα ποσοστά επιβολής για κάποιες υπηρεσίες, υψηλής ε, πυκνότητας εργατικού δυναμικού. Η γυναίκα του του είχε πει ότι μειώσατε το ποσοστό για τον κομωτή μου, αλλά ο κομωτής μου δεν μείωσε τις τιμές του, ούτε και ο δικός μου κομωτής. Και του το ζήτησα. Γιατί δεν το μείωσες? Και η απάντηση του κομιτή ήταν ότι αν δεν είχε υπάρξει μείωση του ε, φόρου θα έπρεπε να αυξήσω το τίμημα της υπηρεσίας μου. Λοιπόν το ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιπτώσεις και για τα εστιατόρια. Υπάρχουν εστιατόρια στο Στρασβούργο που δείχνει πόσο μείωσαν τις τιμές τους. Το λένε αυτό. Δεν παίζει βέβαια απόλυτα ο ελεύθερος ανταγωνισμός, περισσότερο η διαφήμιση. Πάντως σε ορισμένες χώρες δημιουργήθηκαν κάποια θετικά βήματα. Στη Γερμανία το σύστημα είναι εντελώς ανόητο με αποδείξεις κτλ. Αλλά αυτά όλα τα αποφασίζει κυρίαρχα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κάζα και δεν θα πρέπει να ανακατεύουμε τα πάντα και τις απάτες και το ποσοστό επιβολής και τα λοιπά. Εδώ μας ρωτάνε, συμφωνείτε με μια διεύρυνση του μεταβατικού καθεστώτος το οποίο ισχύει. Δεν μας αρέσει το καθεστώς αυτό, αλλά δεν υπάρχει πλειοψηφία για αλλαγή. Θα πρέπει να το δεχτούμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Θα δούμε μέχρι τότε τι άλλο θα σκεφτούμε και να μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι έχουν γίνει αρκετές προτάσεις σχετικά με τους ιδίους πόρους και οι προτάσεις αυτές άπτονται φυσικά του ποσοστού επιβολής ΦΠΑ. Ευχαριστώ. Ασέα. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι θετικές οι προτάσεις ε, του κυρίου Κάζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα τις βοηθήσουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Πράγματι το ΦΠΑ είναι ε, μια επιβάρυνση ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες οι οποίες ακριβώς προέρχονται από έντονη παρουσία εργατικού δυναμικού και δεν υπάρχει διαμεσολάβηση οικονομική και δεν υπάρχουν ε, εξωτερικές πρότεσίλες κτλ. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες αυτές ε, δεν έχουν καμία δυνατότητα να διαφύγουν ή να μειώσουν το ύψος επιβολής της υπηρεσίας, της φορολογίας την οποία υφίστανται οι υπηρεσίες τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να φανταστούμε με διαφορετικούς τρόπους να τους φορολογήσουμε. Δεν ξέρω μήπως, λέει ο κύριος Σικλούνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας μιλήσει λίγο για τα μελλοντικά σχέδια μεταρρύθμισης του ΦΠΑ. Ρακώνει από την Επιτροπή. Να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για μια τεχνική πρόταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει την παράταση για πέντε χρόνια του κατώτερου ποσοστού επιβολής. Δεν πρόκειται τώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μέλλον του ΦΠΑ και για τις νέες στρατηγικές του ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος Σιμέτα το είπε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της ακρόασής του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν παρουσίασε ε, θα παρουσιάσει μάλλον πριν το τέλος του χρόνου ένα πράσινο βιβλίο το οποίο θα καλύψει τα θέματα που περιλαμβάνονται στις τροπολογίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις εσωκοινοτικές συναλλαγές, το πώς θα πρέπει να αντεπιστούν και στο θέμα του ΦΠΑ μεταξύ του οποίου και το θέμα του ποσοστού επιβολής. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν με λίγο ομόλογο και βρίσκω ότι είναι πρόωρο να τροποποιήσουμε την πρόταση αυτή, την ημερομηνία, δηλαδή για το τέλος του 2013. Θα παρουσιαστεί το πράσινο βιβλίο στο τέλος του χρόνου. Θα γίνει αντικείμενο διαβούλευσης για τουλάχιστον έξι μήνες. Θα υπάρξει μετά μια διαβούλευση επίσημη με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επίπεδο νομικής διασφάλισης της διαδικασίας αυτής είναι προτιμότερο να διατηρηθεί η πρόταση του 2015 και όχι του 2013. Είναι νωρίς το 2013. Κύριε Κάζα, να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά όλα τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι. Πράγματι η έκθεση αυτή αναφέρεται σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να συμφωνήσουμε για την χρονική παράταση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια καινούργια πρόταση για τη στρατηγική στον τομέα του ΦΠΑ, προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση και με μας και θα πρέπει εμείς ε, σε κάθε απόφαση που θα ληφθεί να έχουμε πάρει μέρος. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα θα συμφωνήσουμε νομίζω, δεν υπάρχει τόσο φοβερή διαφορά. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι μονίμως σε διαβούλευση με την Επιτροπή μας. το οφείλουμε και στον τομέα τον επιχειρηματικό τον ακούμε τον επιχειρηματικό τομέα και πρέπει να αποφύγουμε να τον επιβαρύνουμε αδικαιολόγητα. μια γιορτή έξω από το κτίριο και έχουμε και καλό κρασί. Μπορείτε να έρθείτε. Από τη Μάλτα. the the chair is biased, so I cannot him. Uh, Εγώ είμαι προκατηλημένος για το κρασί, λέει ο Πρόεδρος. Θα δω τι θα κάνω. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 8η Οκτωβρίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα είναι 26 Οκτωβρίου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει η η την 9η Νοεμβρίου και αν πάνε όλα καλά θα πάμε στην Ολομέλεια είτε του μηνός Νοεμβρίου ή ίσως να γλιστρήσουμε στο Δεκέμβρη. Δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα. Αυτά θα κλείσουμε τη συζήτηση. Αυτή δεν έχουμε άλλα θέματα σήμερα. Αύριο το πρωί στις 9, Θεός να είναι καλά, θα ξεκινήσουμε με το σημείο 6. Α, όχι, με διορθώνει ο γραμματέας. θα έχουμε το πρώτο θέμα, τα ενδιάμεσα μέτρα, το 7 δηλαδή, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο στις 9. Ε, λοιπόν, 10 και μισή ξεκινάμε ψηφοφορίες, μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Thank you